το πρωί, 10 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί και το απόγευμα από τις 3. Η ημερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι καλή νύχτα.